Hezké odpoledne, kolegové. Denní zasedání pokračuje. Vidím, že se hlásí pan Romeva Rueda. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζουμε την απογευματινή σύνοδο. Ο κύριος Ρωμέβα Ρουέδα βλέπω να ζητά το λόγο. Μία πληροφορία που μόλις έμαθα θα ήθελα να σας ανακοινώσω. Εδώ και λίγες εβδομάδες ε, αντιμετωπίζουμε ένα νέο φαινόμενο άνευ προηγουμένου γύρω από μερικές μεγάλες πόλεις της Δυτικής Σαχάρας. Πάνω από 10.000 Σαχαραουίτες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, εκενώνουν τις πόλεις τους ε, και εγκαθίστανται σε σκηνές ε, γύρω από το Αλεγιούν Σμάρα και Μπούστον. Είναι μια νέα μέθοδος διαμαρτυρίας κατά της αβάσταχτης πολιτικής και κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των αυτόχθονων πληθυσμών της Δυτικής Σαχάρας και το λέω αυτό σήμερα γιατί υπάρχει πρόβλημα με τις ε, ε, αιματηρές επεμβάσεις της μαροκινής κυβέρνησης που δυστυχώς αυξάνονται ανησυχητικά. Ζητώ λοιπόν το Ευρωπαϊκό, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει τιμότητα δράσης δεδομένης της νέας κατάστασης. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το σημειώνουμε, αν και δεν ήταν διαδικαστικό, κύριε Ρωμέβα. Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα και η κατάσταση στο Μαρόκο δεν είναι θέμα της απογευματινής συζήτησης, γιατί δεν είναι το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Χθες οριστικοποιήθηκε η σημερινή ημερήσια διάταξη για το απόγευμα. Υπάρχουν καταρχήν ως προς τα χθεσινά πρακτικά αντιρρήσεις. Όχι, οπότε εγκρίνονται και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης.